Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα κάνω πρώτα μια ανακοίνωση. Έλαβα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αιτήσει διορισμού στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος αυτών των διορισμών θα περιληφθεί στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση και αν δεν έχουν υποβληθεί παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, αυτοί οι διορισμοί θα θεωρηθούν ως εγκριθέντες. Τώρα έχουμε την... Τα του Δικού Συμβουλίου Εκοφήν τη 7η Σεπτεμβρίου και τη δηλώση Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Εξ ονόματο του Συμβουλίου θα δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, τον κύριο Ρέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ απλά θα ήθελα να σας πω τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες μας επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σε δύο φακέλους εγκρίνοντας το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την άλλη διαδικασία παρακολούθηση.